Καθυστερήσαμε λίγο διότι πριν ξεκινήσει αυτή η συνεδρίαση της Επιτροπής ε, προπολογισμού είχαμε μία κοινή ε, ε, συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού και Προϋπολογισμού για να ε, συντονίσουμε τη δράση μας σχετικά με τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Τώρα λοιπόν άπαξε τελείωσε εκείνη η υπόθεση μπορούμε να προχωρήσουμε με τον προϋπολογισμό. Σήμερα το απόγευμα, αύριο πρωί και απόγευμα απόγευμα και την πέμπτη το πρωί έχουμε την μακριά συνηθισμένη συνεδρίαση ψηφοφοριών για τις τροπολογίες του προϋπολογισμού αλλά με μία νέα τροπολογία διότι σύμφωνα με την συνθήκη της Λισαβόνας σε κάθε ένα από τα θεσμικά όργανα θα γίνεται μόνο μία ανάγνωση οπότε αυτή η ψηφοφορία είναι ακόμη πιο σημαντική από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα το απόγευμα ε, εξετάζοντας ε, τις ε, δαπάνες της κατηγορίας 5 για τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής. Μετά θα συζητήσουμε το, την έκθεση της Έλγα Τρίπελ για τα υπόλοιπα θέματα και από αύριο το πρωί θα ασχοληθούμε και με τις άλλες κατηγορίες του προϋπολογισμού. Εν τω μεταξύ όπως το γνωρίζουν και τα άλλα μέλη που ήταν στη συνεδρία συγκεκρισμένων των θυρών σήμερα το πρωί πρέπει ακόμη να υπάρξουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των ομάδων για να έχουμε την πλειοψηφία την οποία χρειαζόμαστε. Σήμερα το πρωί συνεδριάσαμε και κλεισμένων των θυρών ώστε οι κατάσκοποι των άλλων ε, οργανισμών να μην ξέρουν τι γίνεται και τι συζητάτε εδώ για λογαριασμό τους. Κατόπιν αυτού θέλω ε, να καλωσορίσω τους νόμιμους εκπροσώπους των άλλων θεσμικών οργάνων και να δώσω αμέσως το λόγο στον Γενικό Διευθυντή Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ως συνηθίζεται ζήτησε να μας παρουσιάσει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορος και σύντομος και καταρχήν θα ήθελα ε, να αναφερθώ εις ε, τις πιστώσεις δεσμεύσεων και επίσης να σας πω ότι ε, η Επιτροπή ε, αξιολογεί τις ε, και εκτιμά τα σχόλια σχετικά με την νεολαία. Επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι σας ενδιαφέρει το 1α και το κεφάλαιο 4 αλλά εμείς θέλουμε να σας πούμε ότι δεν μπορούμε να δεχούμε τροπολογίες που ξεπερνούν τα όρια Δηλαδή σχετικά με το κεφάλαιο 4, ε, εκτός από την Παλαιστίνη θα πρέπει να βρεθούν επιπρόσθετοι πόροι για το Πακιστάν, διότι όπως ξέρετε θα υπάρξει ένα συνέδριο των δωρητών και θα πρέπει να ευρεθεί για την περίοδο μέχρι το 2013 ε, χρηματοδότηση και στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου θα θέλουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων μας. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τα μέλη της Επιτροπής αυτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίοι ε, έχουν αποκαταστήσει ε, τις ε, πιστώσεις πληρωμών διότι το επίπεδο που είχαμε προτείνει σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντικατοπτρίζει ακριβώς τις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον εισηγητή, ο οποίος αποκαθιστά τις περισσότερες πιστώσεις όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ε, ειδικέ. Ε, ε, ε, πρωτοβουλίες που αναφέρονται στα διοικητικά έξοδα των διαφόρων προγραμμάτων διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έκανε την, επέβαλε περιορισμού στον εαυτό της την πρότασή της στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας και γι' αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού ήδη αντί να αυξήσει το προσωπικό της προέβλεπε μία μείνωσή του ελαφρύ. Αλλά αν ε, ε, οι προτάσεις ε, της, του Συμβουλίου διατηρηθούν για το 2011 αυτό θα επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα επιτρέψει ούτε την εφαρμογή των δυνατοτήτων της συνθήκης Λισαβόνας ούτε την διεύρυνση των εντολών μας οπότε πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το κόστος το οποίο προτείνει το Συμβούλιο θα μειώσει το προσωπικό το, το, το, το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 374 ε, υπαλλήλους και 368 συμβασιούχους ε, και ε, είναι δηλαδή μια σημαντική περικοπή. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που αναφέρονται στις διοικητικές πιστώσεις. Θα επανέλθουμε στα σχετικά ε, με την ε, ε, Επιτροπή Συνδιαλλαγής και θα δώσουμε ό,τι πληροφορίες μας ζητηθούν. Θα ήθελα όμως αυτή τη στιγμή να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να ελέγχει και να εξετάζει το προσωπικό της, ενημερώνει συχνά το Κοινοβούλιο και ήδη συνοψίζει ορισμένες θέσεις και από 31 της ε, του προσωπικού στηρίξεως πέσαμε στο 21% το 2010 και θα μειωθεί ακόμη στο 2011. Θέλω να αναφέρω τρία σημεία. Καταρχήν πόσο είναι ανάγκη να περιγράψουμε το πεδίο δράσεως και το, τις πιστώσεις που είναι στα απόθεμα για να μην υπάρξει διακοπή σε ορισμένες υπηρεσίες εις βάρος, εις βάρος πολλών προτεραιοτήτων. Δεύτερον, εάν η η ε, τοποθέτηση σε απόθεμα ε, των μισθών ε, επεκταθεί άλλες, άλλα αποθέματα θα πρέπει να συνοψιστούν εις, το, στη γραμμή των μισθών στη γραμμη χχ χ001 η, η Επιτροπή Επιτροπή δηλαδή απασχολεί ενιαία το προσωπικό και δεν μπορεί να το διαχωρίσει διότι θα είχε πρόβλημα διαχειρίσεως. Και τέλος, ε, μεταξύ της ε, γραμμής των αποθεμάτων και ε, της κατανομής τους υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί εις τα μέτρα του ΕΑΕΣ διότι ορισμένα θέματα δεν μας βρίσκουν σύμφωνους σχετικά με την δημοσιονομική πειθαρχία διότι ε, εσείς ε, έχετε προβλέψει ότι δεν θα υπάρξει κανένα απόθεμα και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει πολύ προσεκτικά τα, τις ε, πιλωτικές δράσεις και ε, τις προκαταρκτικές δράσεις που μας είχατε κοινοποιήσει πριν το καλοκαίρι. Ε, θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί διότι θέλει να υπάρξει συνεργασία για να μπορέσει να υπάρξει μία ρεαλιστική εφαρμογή εφαρμογή των προγραμμάτων τα οποία θα προχωρήσουν σε υλοποίηση. Και τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι πριν τη συνδιαλλαγή θα παρουσιάσουμε τη διορθωτική επιστολή ε, η οποία ενημερώνει τις ανάγκες και το επίπεδο των πιστώσεων γεωργίας και αλληλείας και επίσης ε, μια επεξηγηματική επιστολή θα σας έρθει συντόμως για να εξηγήσουμε ε, τη λειτουργία των τριών οργανισμών χρηματοοικονομικής εποπτείας σύμφωνα με την τελευταία νομοθετική συμφωνία. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις τις οποίες ήθελα να κάνω εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αρχή των εργασιών σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτές τις διευκρινήσεις οι οποίες είναι και σαφείς και σύντομες και ε, προσέξαμε ιδιαιτέρως διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια μεγάλη προσπάθεια εξοικονομήσεως πόρων σε όσο την αφορά για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ε, εξέλιξη του προσωπικού της ε, ε, παρόλη την εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας και σημειώνουμε αυτά που μας είπατε σχετικά με την τεχνική πτυχή των αποθεμάτων για τη χρηματοδότηση των μισθών και πρέπει όντως να φροντίσουμε άπαξ και θα έχουμε λάβει την καταρχήν απόφαση εάν τελικά αποφασίσουμε αυτή την αποθεματοποίηση να υπάρξει ε, μία λογιστική προσαρμογή η οποία να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και όχι γραμμή προς γραμμή και θα το προσέξουμε ε, και οι υπηρεσίες μας το σημειώνουν. Σας ευχαριστούμε διότι ενδεχομένως θα μπορέσετε να απαντήσετε ε, στους εισηγητές ε, για τα πιλωτικά σχέδια και τις προκαταρτικές δράσεις τα οποία συζητάμε ακόμη μεταξύ πολιτικών ομάδων και σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την συνήθεια και για προφανείς λόγους τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα υπάρξει μία διορθωτική επιστολή για τη γεωργία και την αλληλεία και εσύ κατόπιν των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν της αποφάσεως που έλαβε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την λειτουργία των τριών εποπτικών αρχών χρηματοοικονομικών ε, θεμάτων. Οπότε ξεκινούμε την ψηφοφορία. Θα πρέπει καταρχήν να ελέγξουμε ότι είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε. Δηλαδή ότι όλοι έχουμε ε, φέρει από την ε, αίθουσα εργασίας όπου βρισκόμασταν το δελτίο ψηφοφορίας μας, την κάρτα μας. Διότι βλέπουμε ότι ο εισηγητής ή η εισηγήτρια είναι κακή μαθήτρια και την έχει ξεχάσει. Αλλά θα κοιτάξουμε να τη βοηθήσουμε να επανορθώσει. Αυτό που σας προτείνω και θα προχωρώ αργά για να μην υπάρξει σύγχυση και να μπορέσουμε να ψηφίσουμε γνωρίζοντας ακριβώς τι ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αλλά τουλάχιστον να συμφωνούμε για ό,τι ψηφίζουμε. Ας ξεκινήσουμε με, ε, το έγγραφο που έχει ε, το, την ονομασία 4 RAP της 28 Ενάτου 2010, αυτό το έγγραφο που σας δείχνω και ε, το βλέπετε όλοι, το έχετε όλοι μπροστά σας. Εδώ υπάρχουν ορισμένες ψηφοφορίες συνολικές που αναφέρονται σε ορισμένες πολιτικές συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί ή θεωρούνται ότι έχουν επιτευχθεί σε αυτό το στάδιο. Δεν είμαστε ακόμη σύμφωνοι εφόλης της ύλη, αλλά σε ορισμένα σημεία μεταξύ πολιτικών ομάδων έχουμε μία συμφωνία για να ψηφίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Έχετε όλοι αυτό το φυλάδιο μπροστά σας διότι αντιλαμβάνομαι ότι στις δύο τελευταίες γραμμές οι φίλοι μας της σοσιαλιστικής ομάδος δεν είναι σε θέση τώρα να ψηφίσουν τις δύο τελευταίες γραμμές και ζητούν επιπλέον χρόνο για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με τον εισηγητή και τις άλλες ομάδες για να μπορέσουν να συμφωνήσουν. Οι υπόλοιπες γραμμές μπορούν να υποβληθούν σε μία ψηφοφορία. Ναι, ωραία. Λοιπόν, έτσι θα προχωρήσουμε. Πρώτη ψηφοφορία τώρα, οι πολιτικές προτεραιότητες, ε, τα, οι οριζόντιες τροπολογίες του εισηγητή για την νεολαία, την παιδεία και την κινητικότητα μπορούμε να ψηφίσουμε ε, συνολικά. Τότε όλη τη σελίδα αυτή την υποβάλλω προς ψήφιση ε, μαζί. Ποιος είναι υπέρ κατά, δύο κατά, αποχές, καμία αποχή και ο συντονιστής του ΕΛΚ κατάλαβε τώρα τι ψηφίζουμε. Αλλά χαμογελάει, άρα δεν είναι αρνητικός. Μπορούμε λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε στην οριζόντια προσέγγιση του εισηγητή για τις υπηρεσίες, δηλαδή τη σελίδα 2 και 3. με την συμφωνία της Γιούτα Χάουκ, της ειδική εισηγήτριάς μας, ψηφίζεται ολόκληρο ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δύο κατά, αποχές, μία αποχή. άρα υπερψηφίστηκε, αλλά η Αν θέλει να κάνει μία δήλωση. Και εμείς ψηφίσαμε τα 4 εκατομμύρια υπέρ των συμφερόντων της Ελίας. Αντιλαμβάνομαι ότι όσα αναφέρεται ε, στην ε, υπηρεσία αλληλείας θα υπάρχει χωριστή ψηφοφορία όταν θα φτάσει η στιγμή. Συμφωνεί ο εισηγητής αλλά θα υπάρξει χωριστή ψηφοφορία ε, προς τιμήν της Αν Γένσεν και της ομάδας της για να μπορεί να πει ότι θα υπήρχε μία συγκεκριμένη ψηφοφορία για, αυτή την, για αυτό τον οργανισμό οργανισμό και όχι ε, για, μαζί με, τις, με τους άλλους οργανισμούς συλλήβδιν ακόμη και αν πρόκειται για την επιστημιστική ε, ασφάλεια και διατροφική ασφάλεια θα έχει μία ειδική αντιμετώπιση αλληλεία. Τώρα ερχόμαστε στις σελίδες 4 και 5 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές μία αποχή. Δύο κατά και μία ψοχή, αποχή, βρία αποδοχή, άρα και αυτή η προσέγγιση υιοθετείται. Τώρα έχουμε την οριζόντια τροπολογία του εισηγητή σχετικά με ε, το 1,85% ε, αύξηση ε, των μισθών που πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι οι γραμμές από τη σελίδα 6 έως 9, είναι η ίδια υπηρεσία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος είναι υπέρ, αλλά αναφέρεται σε διάφορους τομείς. Ποιος είναι υπέρ και πάλι. Το ΕΛΚ είναι κατά. Ας κάνουμε τότε ηλεκτρονική ψηφοφορία διότι θα μας βοηθήσει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, το, την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ωραία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Παρακαλώ την γραμματεία να εξασφαλίσει ότι καμία πολιτική ομάδα δεν έχει υπεράριθμους. Ο εισηγητής όμως είναι υπέρ. Ωραία. Λίγη ψηφοφορία. 22 υπέρ, 15 κατά 23 υπέρ, 15 κατά, άρα αυτή η τροπολογία υιοθετείται, πρόκειται για την οριζόντια τροπολογία για τη διαχείριση των μισθών και των ε, συντάξεων. Αυτό εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα θεσμικά όργανα. Μήπως κάποιος ζητά να γίνει η ίδια ψηφοφορία και για τα άλλα θεσμικά όργανα, διότι κανονικά πρέπει να υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση ασχέτως του θεσμικού οργάνου, εφόσον όλες οι, ε, όλα τα θεσμικά όργανα έχουν εναχθεί. Εφόσον συμφωνείτε λοιπόν, ισχύει η ψηφοφορία για όλα τα θεσμικά όργανα. Και τώρα φτάνουμε σελίδα 10 η οριζόντια προσέγγιση του εισηγητή για το κεφάλαιο 5 εκτός αυτό το σημείο το οποίο μόλις ρυθμίσαμε της προσαρμογής ε, των μισθών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ένας κατά. Αποχές. Μία αποχή. βρία λοιπόν συνένεση και υιοθετείται και τελευταία ψηφοφορία η οριζόντια ε, ε, τροπολογία για τις μελέτες σελίδα 11 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές μία αποχή και έτσι αποφασίζουμε και νομίζω ότι προχωρήσαμε πολύ. Λοιπόν, Άπαξ ε, και έχουμε συμφωνήσει σε αυτές τις καταρχήν τροπολογίες μπορούμε να ξεκινήσουμε το, ε, την εξέταση της κατηγορίας 5. Οπότε παρακαλώ να πάρετε ε, το φυλάδιο με όλες τις τροπολογίες. Εσείς δεν έχετε ίσως τον τοσχέ απ' έξω, αλλά είναι το ίδιο. Bon. Euh, λοιπόν, διοίκηση. Ε, όλοι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος ε, κείμενο, στο αγγλικό κείμενο, είναι το 163 Δεν ξέρω αν εσείς με καταλαβαίνετε, εγώ όμως με καταλαβαίνω. Αν κάποιος έχει ε, δυσκολίες... Ο κύριος Κολίνο έχει δυσκολίες. Η σελίδα 163, η Επιτροπή χωρίς τις συντάξεις. Ε, η τροπολογία 4762 του κυρίου Ερενχάουζερ καλύπτεται όπως και το 46 66 ε, ε, του κυρίου Ερενχάουζερ αλλά η 46-65 δεν καλύπτεται ποιος, ο, ποιος είναι υπέρ ευχαριστώ άρα απορρίπτεται στο 416 της ΕΚΟΝ. Ποιος είναι υπέρ, ο εισηγητής είναι υπέρ. Κατά. Άρα υιοθετείτε. Το 42 21 της κυρίας Βαλζάνη ε, έχει καλυφθεί και τώρα Ψηφίζουμε το 63 Τις παρατηρήσεις δηλαδή. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Απορρίπτεται. Οι τροπολογίες δηλαδή αυτές απορρίπτονται και για όσους έχουν το ίδιο τετράδιο γυρίζουμε σελίδα. Δεν ε, ψηφίζουμε το 4367 για την πιλωτικό πρόγραμμα και ακόμη δεν έχουμε συμφωνήσει με τις ομάδες για τα πιλωτικά θέματα. Η τροπολογία Ερενχάουζερ έχει καλυφθεί και το 4605 το 4532 του κυρίου Ερεν Χάουζερ. ποιος είναι υπέρ κατά ευχαριστώ Οι, οι τρεις ε, επόμενες ε, τροπολογίες ε, ε, καλύπτονται. Πρέπει όμως να ψηφίσουμε την 4531 του κυρίου Ερενχάουζερ. Ο, ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Ένας υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι επόμενες τρεις τροπολογίες καλύπτονται, το 47-45, το 45-98 και το 467 επίσης καλύπτονται. Αλλά πρέπει να ψηφίσουμε το 45-50 του κυρίου Έρενχάουζερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όλες οι τροπολογίες της σελίδος 166 έχουν καλυφθεί. Όχι. Η συγγήτρια, ναι, και εγώ έλεγα ότι παρά ήταν αισιόδοξη η δήλωσή μου. Τι έχει να μας πει η συγγήτρια επ' αυτού. Ο κύριος Χάρτουγκ έχει κάποιο πρόβλημα. Είμαστε σελίδα 166. στο επάνω μέρος της σελίδας η γραμμή 050101 έξοδα σε σχέση με το προσωπικό σε ενεργή ε, δράση στη γεωργία και στην ανάπτυξη της υπαίθρου και τη σχετική πολιτική. Η συντονία. Όλες οι τροπολογίες αυτές καλύπτονται εκτός από τις, τα αποθέματα και τις συνθήκες αποθεματοποιήσετος και εγώ είμαι ενάντια σε αυτές τις παρατηρήσεις και σε αυτό το απόθεμα. Ωραία. Λοιπόν, στη σελίδα 166 όλα καλύπτονται εκτός όπως μου λέει ο εισηγητής η τροπολογία 406 η οποία αναφέρεται σε αποθεματοποίηση και σε ένα σχόλιο σχετικά με την αποθεματοποίηση. Οπότε, για τις άλλες τροπολογίες δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε, Ποιος είναι υπέρ της ε, ε, ε, αποθεματοποιήσεως είναι για την γνωστή υπόθεση του καπνού και βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί εχθροί του καπνού. Ψηφίζουμε για τον καπνό. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας αυτής. Ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λίγη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λίγη. 22 υπέρ 15 κατά η τροπολογία υιοθετείται οπότε κανείς πια δεν πρέπει να, να καπνίζει μέσα στην αίθουσα. Τουλάχιστον δεν θα επιδοτούμε πλέον τους καπνιστές. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην επόμενη σελίδα, στην 167 όπου έχουμε την ε, τροπολογία 4137 του κυρίου Χάρτονγκ. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Ο κύριος Αρτόν και κανείς άλλος. Ποιος είναι κατά. Όλοι. Ε, αποχές καμία αποχή, άρα απορρίπτεται. Τώρα έχουμε το 45-49 του κυρίου Έρενχάουζε. Ο εισηγητής είναι κατά. Ε, ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. Το 46.00 καλύπτεται, το 45.48 πρέπει να υποβληθεί σε ψηφοφορία, εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Οι τρεις άλλες τροπολογίες μέχρι το τέλος της σελίδας 4142, 41-42, 47-43, 41-42. Γυρίζω σελίδα και γυρίζω στο, τη σελίδα στο Other Management Expenditure το 4142-4601 καλυπτεται και θέτουμε προς ψηφοφορία στη 45.47 του κυρίου Ερεν Χάουζερ. Ποιος είναι υπέρ, ο, ο εισηγητής είναι κατά, κατά, απορρίπτεται. Το 47-40 καλύπτεται, το 46-02 καλύπτεται, ψηφίζουμε τη 45-46. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 41-44 καλύπτεται, 46-03 καλύπτεται, ψηφίζουμε τη 45-45. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. 41-46 καλύπτεται, 47-41 καλύπτεται, 45-3 καλύπτεται, 45-44 του κυρίου Ερενχάουζερ πάλι ψηφίζεται ποιος είναι Κατά. για να διευκολυνθεί η εργασία μας βλέπω ότι ο κύριος Ερενχάουζερ στο κεφάλαιο 5 έχει καταθέσει τροπολογίες ε, σε όλες τις γραμμές για να μειωθούν κατά 10%. Σε 20 ψηφοφορίες βλέπουμε το ποσοστό είναι το ίδιο. Οπότε θα έλεγα ότι όποτε υπάρχουν τέτοιες τροπολογίες στο κεφάλαιο 5, θα δούμε για τα άλλα, θα θεωρήσουμε ότι ισχύουν οι ίδιες ε, πλειοψηφίες εκτός και αν κάποιος αμφισβητήσει και μου το πει. Οπότε το 45-94 απορρίπτεται, το 45-43 ε, ε, ε, η ίδια, ψηφο, η ίδια πλειοψηφία, 47-42 καλύπτεται, 45-95 καλύπτεται, 45-42 η ίδια πλειοψηφία, 47-38 καλύπτεται, 45-96 καλύπτεται, 45-41 η ίδια πλειοψηφία, 2-83 καλύπτεται, είναι η Επιτροπή Πολιτισμού που είναι πολύ ευτυχής όπως και για το 284 που καλύπτεται. Το ίδιο και για το 4597 και το 285 για την Επιτροπή Πολιτισμού. 45-40. Κύριος Ερενχάουζερ, η ίδια πλειοψηφία. Στην επόμενη σελίδα 172. Όλες οι τροπολογίες έχουν καλυφθεί εκτός από το 3502 όχι έχει καλυφθεί και αυτό άρα όλη η επόμενη ε, σελίδα 172 έχει καλυφθεί με τον ίδιο τρόπο όλη η σελίδα 173 εκτός από τις δύο τελευταίες γραμμές. Βρίσκουμε λοιπόν στην τροπολογία 535, πρώτη τελευταία τροπολογία που έχει κατατεθεί από το ΕΛΚ, που έχει μία επιφύλαξη σχετικά με την πληροφόρηση. Ο εισηγητής είναι υπέρ της ε, επιφύλαξη αυτής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ αποχές η πλειοψηφία είναι υπέρ, άρα η επιφύλαξη αυτή υιοθετείται. Στο 4530, στο κάτω μέρος της σελίδας, έχουμε πάλι την ίδια πλειοψηφία για τις τροπολογίες μειώσεως κατά 10% του κυρίου Έρεν Χάουζερ. Το ίδιο συμβαίνει και με το 4631. Αντιθέτως, η 627 είναι μία τροπολογία των φιλελευθέρων της ομάδας των φιλελευθέρων που κατακρίνει την ε, χρήση η οποία έχει γίνει στο παρελθόν. Είναι δηλαδή μία τροπολογία επί των σχολείων. Ο εισηγητής θα συζητάει το λόγο. μια επεξήγηση μια αρχή γιατί υπάρχει μια σειρά τροπολογιών για την παρατήρηση, αξιολόγηση αυτού του κονδυλίου και συνιστώ να καταψηφιστούν. Ωστόσο όμως σημειώνω πολύ καλά το μήνυμα διότι πιστεύω ότι δεν είναι εδώ η θέση να εισαχθεί αυτό το μήνυμα. Όμως για το ψήφισμα σίγουρα είναι μια επιλογή να συμπεριληφθεί εκεί τροπολογία για το ψήφισμα με αυτό το κρίσιμο μήνυμα, τότε θα είμαι υπέρ. Όχι όμω ω σχόλια σε αυτό το κονδύλιο. Γι' αυτό η σύστασή μου είναι να καταψηφιστούν εδώ. Ευχαριστώ. Δηλαδή η ιδέα του εισηγητή είναι ε, να σημειώσει την ε, κριτική η οποία εξασκείται και να την τονίσει εις ε, το ψήφισμα το οποίο θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια μαζί με τις τροπολογίες μας. Θέλει μήπως η ομάδα των φιλελευθέρων να αποσύρει αυτή την τροπολογία υπέρ των σχολείων του εισηγητή, κυρία Γέντσεν. Ουσιαστικά δεν αποσύραμε αυτή την τροπολογία διότι για τη χρήση ακριβώς των χρημάτων θεωρούμε ότι ισχύει ακόμα, είναι ισχυρή. Υποβάλλω αυτή την τροπολογία προς ψήφιση. Ο είναι κατά. Ποιος είναι Κατά. Αποχές. Τα δύο μαμούθη λοιπόν απορρίπτουν αυτή την τροπολογία. Μία άλλη τροπολογία και πάλι της ομάδας του κυρίου Αλβάρο είναι ταυτόσιμη αλλά για μία άλλη γραμμή του προπολογισμού. Καλύπτεται και αυτή. Άρα δεν χρειάζεται η επόμενη τροπολογία να ε, ψηφιστεί. Θέλετε να ξαναψηφίσουμε. Κυρία εισηγήτρια. Πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσουμε την 4661 του κυρίου Έρενχάουζεν. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε έτσι χωρίς να υπάρξει κάποιο σχόλιο. Je vous demande pardon. Ε, Με συγχωρείτε. Καταρχήν θα ψηφίσουμε την 4353 ε, που είναι στο ίδιο πνεύμα με την 627 την οποία μόλις ψηφίσαμε και μετά θα ασχοληθούμε με τη 4631. Ε, ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ της 4353. Κατά. Αποχές και πάλι ίδια πλειοψηφία όπως και στην 627. 4631 του κυρίου Έρενχάουζεν. Είναι ε, μία τροπολογία για μείωση πιστώσεων αλλά δεν είναι συνηθισμένη όπως σε άλλες γραμμές όπου ζητά 10% εδώ προτείνει διαφορετική ε, μείωση. Ο εισηγητής είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, μία αποχή απορρίπτεται συνεχίζουμε και φτάνουμε στα πιλωτικά σχέδια. Το 281 δεν θα το ψηφίσουμε διότι δεν υπάρχει συμφωνία για τα πιλωτικά προγράμματα. Περνάμε στο 309 το οποίο υποβάλλω προς ψήφιση, ο εισηγητής είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά, γιατί νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή πολιτική διαφωνία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Υπάρχει ένα σοσιαλιστής παραπάνω. Αυτό είναι κακό. Πρέπει να σκοτώσουμε έναν σοσιαλιστή. Κάποιος αυτοκτόνησε. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι σαφής 30 κατά, 12 υπέρ, εκ των οποίων ένα αφιλεγόμενος σοσιαλιστής, άρα απορρίπτεται. Το 663 ε, καλύφθηκε, το 4228 καλύφθηκε, στην επόμενη σελίδα όλα έχουν καλυφθεί ή όχι. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η 405 για το καπνό καλύφθηκε από την προηγούμενη ψηφοφορία. Ε, είναι διαφορετικά. Είναι πάλι καπνός, αλλά για διαφορετική χρήση του καπνού. Αυτό... Από την Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι το δεύτερο ήμιση του αποθεματικού για την ίδια εκστρατεία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να απαντήσει τι γίνεται. Καλύπτεται με την πρώτη ψηφοφορία μας ουσιαστικά αυτό. Κατάλαβα. Δηλαδή, η 47-39 έχει καλυφθεί, το 247 έχει καλυφθεί, το 45 πρέπει να ψηφιστεί, ο εισηγητής είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. Και πάλι ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ε, τροπολογία 405 και παρακαλώ τους σοσιαλιστές να μην είναι υπεράριθμοι γιατί δεν θα κερδίσουν έτσι. Ψηφίσατε όλοι. Ψήφισαν 41, άρα σωστά. 15 είναι υπέρ, 25 κατά, άρα απορρίπτεται. Το, η 423, η αποθεματοποίηση πιστώσεων για την ΕΦΣΑ. Ποιος είναι ε, υπέρ. Κατά. Οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι και ο ο κύριος Χάρτουγκ. Άρα η 423 υιοθετείται. Το 242 έχει καλυφθεί, το 4591 έχει καλυφθεί, το 4529 είναι αυτό το οποίο ονομάζω τη ίδια ε, πλειοψηφία, έχει καλυφθεί και το 249. Στην επόμενη σελίδα έχει καλυφθεί, 46-90 ίδια ψηφοφορία. Το, οι τρει επόμενε Ερενχάουζερ καλύπτονται ή όχι, όχι, με συγχωρείτε, προχώρησα πάρα πολύ γρήγορα. Επανερχόμαστε στην αρχή της σελίδας 176. Η τροπολογία 194 της Επιτροπής Ελευθεριών περιλαμβάνει ένα σχόλιο και ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ο κύριος Χάρτουγκ και μία αποχή για την ελευθερία. Άρα το σχόλιο αυτό υιοθετήθηκε. 45-38 του κυρίου Έρενχάουζερ η ίδια πλειοψηφία το 47-60 έχει καλυφθεί, το 42-35 τη Ίγκεπ Γκρέσλε. Υπάρχει ε, ε, μία, αναφέρεται μία, σε ένα απόθεμα, ο εισηγητής είναι κατά, αλλά η Ίγκε είναι υπέρ. Δεν είναι όμως εδώ, άρα αυτό μας διευκολύνει. Ποιος είναι κατά. Ο κύριος Σούρια. Καλύπτεται από τροπολογία του ΕΛΚ σύμφωνα με τη δική μας εκτίμηση. Ναι, αλλά δεν έχουμε ψηφίσει ακόμη. Εφόσον δεν είναι εδώ δεν μπορούμε ε, να την εκπροσωπήσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν. Και ξαναξεκινώ την ψηφοφορία σχετικά με τη 42-35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποσύρεται εάν καλύπτεται από μία άλλη τροπολογία του ΕΛΚ θα την ψηφίσουμε στη συνέχεια. Ο κύριος Έρενχάουζερ 4759 και πάλι ήδη ε, πλειοψηφία, άρα δεν ψηφίζεται και η 519 είναι το απόθεμα του ΕΛΚ και ο εισηγητής με ζητά το λόγο. Ευχαριστώ. Συνιστώ να υπερψηφιστεί. Όμως πρέπει να προειδοποιήσω τα μέλη ότι τα ποσά θα πρέπει να προσαρμοστούν, διότι είναι μέρος, τμήμα της οριζόντιας τροπολογίας μας. Προτείνω να ψηφίσουμε για τα σχόλια και μετά για το ποσό που θα εγγραφεί. Ιστερότερα να ψηφίσουμε για το ποσό. Donc, on vote ή να προσαρμοστεί με τεχνικό χαρακτήρα. Εντάξει, δική σας επιλογή. Λοιπόν, αυτή είναι η τάξη μεγέθους, αλλά ο αριθμός θα διευκρινιστεί κατόπιν των αναγκαίων τεχνικών προσαρμογών. Ο εισηγητής με αυτή την ε, ε, απόφαση είναι υπέρ. Ποιος άλλος είναι υπέρ, κατά. Ας ψηφίσουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος. όλοι ψηφίσαν θαυμάσια. 20 υπέρ, 20 κατά, άρα απορρίπτεται. Α, 21, με συγχωρείτε, 21. Και δεν έχουμε υπερβολικούς ο, του ΕΛΚ εδώ. Ελκατζίδες. Βέβαια α, δεν ξέρουμε, υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι ε, εμφανίζονται από το πουθενά. Άρα το 42 ο 36 της κυρίας ε, Γκρέσλε, ο εισηγητής ε, είναι αντίθετος, ποιος είναι υπέρ κανείς, κατά όλος ο κόσμος, αποχές ορισμένες, άρα απορρίπτεται. Το 45-89 πάλι η ίδια πλειοψηφία του κυρίου Ερενχάουζερ, το ίδιο και το 45-88 αλλά μου λένε ότι το 45-28 είναι διαφορετικό. Άρα ψηφίζουμε τη 45-28, ο είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η ε, 47-58 ε, και 47-57 καλύφθηκε όπως και η 4586 και η 4587 στην επόμενη σελίδα. Η 4527 είναι ίδια πλειοψηφία. Οι τρεις επόμενες τροπολογίες του κυρίου Έρεν Χάουζερ μέχρι το κάτω μέρος της σελίδας 178 καλύπτονται με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο ισχύει για όλη τη σελίδα 179 τις οποίες οι τροπολογίες καρύπτονται εκτός από την 4526 που είναι ε, ε, σαν ε, τα άλλα της μειώσεως του 10% στο οποίο η πλειοψηφία είναι αντίθετη. Φτάνουμε τώρα στο 45 στην επόμενη σελίδα 181 και όλες οι προηγούμενες καλύπτονται, πρόκειται για τις τροπολογίες Χάουζερ για 10%. Δηλαδή ακόμη και το 31-25 καλύπτεται κυρία εισηγήτρια. Εντάξει. Προχωράμε λοιπόν σε σελίδα 181. Η 47-52 καλύπτεται. Η 34 αναφέρεται σε μία μεταφορά και αποθεματοποίηση της κυρίας Γκρέσλε. Λοιπόν, το ΕΛΚ μου ζητά να ψηφίσουμε πρώτα την 514 πριν από τη 42-34, διότι το ΕΛΚ είναι υπέρ της 514, ενώ ο εισηγητής είναι κατά τη 42-34. Κάποιος αντιτίθεται σε αυτή την αναστροφή, οπότε καταρχήν ψηφίζουμε την τροπολογία 514 του ΕΛΚ και αντιλαμβάνουμε ότι ο εισηγητές ε, είναι θετικός. Ε, δεν ξέρω εάν ε, έχω αντιληφθεί σωστά. είναι ένα τεχνικό θέμα για την ψηφοφορία, διότι αν κατάλαβα καλά υπάρχει ε, μία κατάταξη σύμφωνα με τα ποσά και το ποσά είναι τα ίδια. Πιστεύω λοιπόν ότι η τροπολογία 517 του ΕΛΚ αν ψηφιστεί καλύπτει και την προηγούμενη. Αλλά μπορούμε να ψηφίσουμε πρώτα τις πρώτες δύο και μετά να αφήσουμε την τρίτη. Δεν είναι όμως η σωστή κατανομή έτσι. Κυρία Συγγήτρια, τι προτιμάτε να ψηφίσουμε την 42-34 πρώτη ή την 514 να ψηφίσουμε πρώτα την 517 και κατά τη γνώμη μου τα άλλα καταπίπτουν. Ωραία. Αρχίζουμε με την 517. Χωρίς νούμερα. Είναι αποθεματικό. Λεπτομερής αύξηση 2011. Ψηφίζουμε την 517. Εισηγήτρια υπέρ. Το ΕΛΚ επίσης υπέρ κατά πλειοψηφία υπέρ. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 517 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε γρήγορα παρακαλώ. Δύο λοιπόν, δύο κοιμώνται φαίνεται. Τόσο χειρότερο για αυτούς. Πέρας. 22 υπέρ. Εγκρίνεται. Η 42-34 καταπίπτει. Υπάρχει ένα στοιχείο στην 517 που αφορά μεταφορά. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε χωριστά. Εγώ είμαι κατά. Πρέπει να ψηφίσουμε όμως. 42-34 καταρχήν. Πριν έρθουμε στην 514, η 42-34, το είπα και πριν κύριε Πρόεδρε, έπρεπε να ψηφίσαμε αντίστροφα. Πρώτα την 5-1-7, με πάση περιπτώσει, δεδομένη τη κατάσταση, προτείνω να ψηφίζουμε την 514 για τη μεταφορά και μετά η 42-34 καταπίπτει αν η 514 ψηφιστεί. Η συγγήτρια είναι κατά της 514 και ψηφίζουμε υπέρ ηλεκτρονικά. Η συγκεκριμένη είναι κατά 514. Το ΕΛΚ τι κάνει. Θέλω κι εγώ να ψηφίσω. Τι λέει το ΕΛΚ. Τι μου λέει. Πέρας. 15 υπέρ 23 κατά απορρίπτεται. Άρα θα ψηφίσουμε την 42-34. Δεν καταπίπτει. Κύριε Πρόεδρε, το ποσό καταπίπτει, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε μόνο το παθηματικό. Ψηφίζουμε τη 42-34, όχι το νούμερο, αλλά το να μπει στο αποθεματικό. Η συγγήτρα είναι κατά. Είναι κανείς υπέρ. Κανένας. Α, η κυρία Ολμάγερ. Κατά. Πολλοί είναι κατά. Αποχές. Με μεγάλη κακή απορρίφθηκε αυτή η τροπολογία. Για τους μισθούς τώρα. 31, 25, 7, 82 καλύπτονται. Special Advisors. Special Advisors. Κάτι θέλει να μας πει η Κομισιόν για τους ειδικούς συμβούλους. 42-30. Κύριε Γενική, έχετε το λόγο. Θα σας πληροφορούμε συνεχώς για τον κατάλογο αυτών των συμβούλων. Σας το λέω, σας το δηλώνω. James Ellis. Επειδή δεν είναι εδώ η είμαι υπέρ αυτής της τροπολογίας, το τονίζω, χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες. Ωραία θα ψηφιστεί η τροπολογία 42-30 υπέρ, η συγκίτρια κατά. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 512 είναι ταυτόσιμη ή όχι. Καταπίπτει. 45-80 η ίδια πλειοψηφία απορρίπτει. «513» για το αποθεματικό Η είναι υπέρ. Υπέρ 513. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 42-32 καλύπτεται, καταπίπτει δηλαδή. 45-37 απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. Οι άλλε τρει τη σελίδα, πειραματικά προγράμματα, δεν τι ψηφίζουμε. 47-36 καλύπτεται. 42-29. Η συγκέντρια είναι κατά. Ψηφίζουμε. Κανείς κατά. Ευχαριστώ. αποχέ απορρίπτεται. 518 και αυτή η αποθυματικό ΕΛΚ εισηγήτρια υπέρ κατά οι σοσιαλιστές αλλά είναι κάπως απομονωμένοι χάνουν εγκρίνεται αυτή η τροπολογία 45-79 καλύπτεται Υπάρχει πλειοψηφία που την απορρίπτει και οι άλλες δύο τις 183 σελίδες καλύπτονται. Γυρίζω σελίδα. Μια τροπολογία της Συντόνια που καλύπτεται, όλα καλύπτονται με την 46-39 του κυρία Χάιζερ, που δεν είναι συνήθις τροπολογία, είναι να μπει στο αποθηματικό του κόστους των κτηρίων η συγγήτρια. Κατά τη 46-39 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η επόμενη καλύπτεται. 46, 40, 46, 57 όπως και 46-38 και 46-53 είναι συνήθεις τροπολογίες, η πλειοψηφία είναι κατά. καλυπτονται καλύπτονται. 46-54-46-55 46-55-46-54 Έρεν υπάρχει μείωση του ποσού αλλά μπαίνει στο αποθηματικό. Λίγο διαφορετική τροπολογία. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Ας αρχίσουμε τη 4654. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Το ίδιο και η επόμενη. 515. ΕΛΚ. Η συγγήτρια κατά υπέρ του ΕΛΚ. Και ο Τζέιμς κατά όλοι οι άλλοι. Αποχές πλειοψηφία κατά. 42-31 καλύπτεται. Ναι. όλη η υπόλοιπη σελίδα. Και η σελίδα 187 όλη καλύπτεται. Η σελίδα 188 στα αγγλικά πάντα Brussels 3, Brussels 4 σαν ονόματα αυτοκρατόρων ακούγονται αυτά, καλύπτονται. Η επόμενη σελίδα, η 189 στα αγγλικά, Λουξεμβούργ 1, Λουξεμβούργο 2 καλύπτονται πλήρω. Η 190 Μόλ. Frankfurt am Καλύπτονται και αυτά. Καλσρούε. Η Συντόνια έχει προφορική τροπολογία και το Είναι μια προφορική τροποποίηση στην 2601-5123 Ευρωπαϊκό Σχολείο στην Καλσρούη. Θα ήθελα να συστήσω να υπερψηφιστεί η τροπολογία 4166. Το ποσό όμως είναι λανθασμένο. Το σωστό ποσό, μη γελάσετε, είναι 14.991 ευρώ. Και αυτό επειδή, επειδή The figure... Μπορείτε να επαναλάβετε το ποσό. Το ποσό είναι 14.991 ευρώ. And not 15. not... Όχι 15 λέει ο πρόεδρος 15.000. Και αυτό γιατί, διότι είχαμε οριζόντια προτεραιότητα ως προτεραιότητα και είχαν συμπεριληφθεί τα ευρωπαϊκά σχολεία. Υπάρχει μια διαφορά. Είναι όμως σημαντικό αυτό το θέμα για αυτό το σχολείο ακούγεται περισσότερο αυτό το ποσό, έχει όμως πρακτικές επιπτώσεις για αυτούς τους μαθητές. Donc on a connu on a connu Riemann Είχαμε Θαλής, Ρίμαν και Λομπαζεύσκη από τη χώρα της, τώρα θα γνωρίζουμε και τη Σιντόνια στη γεωμετρία. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία. 35 υπέρ, γιατί την σε αυτή η αριθμητική. Κατά, αποχές, ευχαριστώ πολύ, εγκρίθηκε. Το υπόλοιπο της Καλστρούε και του Μονάχου εγκρίνονται, όλη η υπόλοιπη σελίδα δηλαδή. Γυρίζω σελίδα. Με εξωτικά ευαινόματα μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Αλικάντε, καλύπτεται Βαρέζε, καλύπτεται Μπέργεν, καλύπτεται Κιόλαμ, καλύπτεται... Αυτά είναι όλα παιδιά της Γιούτα EU contribution to the type 2 European schools καλύπτεται. Όταν όμως έρθουμε στις δαπάνες για το προσωπικό συνεργή υπηρεσία, 47-35 καλύπτεται, αλλά η 42-38 και η 5-16, δύο τροπολογίες για το αποθηματικό, συντόνια έχει το λόγο. Μια ιστορία όπως και πριν αυτή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 Il y a une opposition socialiste libéraux, voilà, mais qui n'est pas majoritaire. Abstention et M. Hartung. Abstention, pas d'abstention, donc il y a une majorité en faveur de cet amendement. Il est adopté, donc le 42-38 tombe, false, ok. 42-38 καταπίπτει. Και περνάμε στην επόμενη τροπολογία να μπει σε επαθηματικό το προσωπικό του Γενικού Γραμματέα ο οποίο έφυγε, έφυγε αυτή τη στιγμή από την αίθουσα, 42-37. Η συγγήτρια είναι κατά υπέρ, κατά, αποχές, με μία ψήφο διαφορά απορρίπτεται. Μπορεί να ξαναγυρίσει ο Γενικός Διευθυντής στην αίθουσα αν θέλει. Δεν θεωρείται περισσότερο να πια. Επόμενη σελίδα. Όλα καλύπτονται Η Συντόνια θέλει το λόγο η τροπολογία Γκάγερ 4305. Δεν ξέρουμε γιατί, ούτε και η ίδια φαίνεται να ξέρει γιατί, αλλά θέλει να μιλήσει. Κάνω λάθος. 4305. Γκάγερ, ο οποίος είναι παρόν. Η Γιούτα, ξέρει, είναι εκπρόσωπος και του κυρίου Γκάγερ και της Συντόνια. Θα μιλήσει για λόγο τους. Είναι τεχνικό σφάλμα αυτό. Αυτό που θέλουμε εκεί είναι τα επιχειρήματα, η αιτιολόγηση να είναι σχόλια. Justifications as remarks έτσι να ψηφιστούν. Αυτό είναι όλο. Κατά τα άλλα παραμένει ως έχει. Κύριε Γκάγερ, συμφωνείτε με την ερμηνεία αυτή. Ναι, ωραία. Αυτό ήθελα να πει και η Συντόνια λοιπόν. Η Συντόνια ξανά έχει το λόγο. Ουσιαστικά δηλαδή λέμε ότι το ποσό καλύπτεται, αλλά θεωρείται ότι τα σχόλια θα, περάσουν, θα πρέπει να περάσουν με μορφή τροπολογίας εγώ είμαι, να ψηφίσουμε, είμαι υπέρ του να ψηφίσουμε κατά. Είμαι κατά. Πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι δύο επόμενες του κυρίου Έρενχάουζερ καλύπτονται. Οι 45-35 ίδια, ίδια πλειοψηφία. Οι άλλε δύο καλύπτονται. Γυρίζω σελίδα στο κείμενό μου. 45-34 ίδια πλειοψηφία. Είμαστε στην 196 του αγγλικού κειμένου, του αγγλικού κειμένου πάντα, όχι στις άλλες γλώσσες. Είμαστε στην 20, γραμμή 28-01-03. 01 Τροπολογία 34 καλύπτεται. 42 42.33 μεταφορά και αποθεματικό. Η συγγήτρια. Έχω να πω κάτι για την γραμμή 29-01-01. Η 34-33 συνδυάζεται με την τροπολογία που, ψηφίσαμε ήδη για τη μεταφορά και καταψηφίσαμε ήδη. Ουσιαστικά καλύπτεται, γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα πιστεύω. Και έτσι πιστεύω η 5-1-4 καταπίπτει και αυτή. Donc, vous voulez dire que... Δηλαδή ουσιαστικά μας λέτε ότι η 42-33 ήδη ψηφίστηκε, καταψηφίστηκε μάλιστα, και η 514 επίσης. Άρα δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Ναι, αυτή είναι η απόψη μου, λέει η συγκέντρωση. Δεν ξέρω αν η ομάδα μου συμφωνεί. Η κυρία Χάουκ μου λέει για την 514 υπάρχουν σχόλια. Remarks. Το ΕΛΚ τι λέει για την 514. Καρίγκα. Να ψηφίσουμε και είναι υπέρ του σχολείου. Bon. Donc c'est uniquement le commentaire. Ψηφίζουμε λοιπόν μόνο το σχόλιο της 514. Bon, alors on me dit qu'il n'y a pas de commentaire sur 514. Εδώ μου λένε οι συμβουλοί μου ότι δεν υπάρχουν σχόλια για το 514. Να ψηφίσουμε το 0, αν θέλετε, να το ψηφίσουμε. Αλλά το μηδέν, πάνω στο μηδέν, πώς να το επηρεάσουμε, το τίποτα. Πάση περιπτώσει, ψηφίζουμε. Για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Οι άλλες δύο τροπολογίες μετά με την ίδια πλειοψηφία καλύπτονται. Περνάμε στη σελίδα 197 την Αγγλική. Εδώ όλα καλύπτονται όλη η σελίδα temporary allowances, pensions of former members και για τους επιβιώσαντες συζύγους και εξαρτώμενα μέλη, ε, επιδόματα για το προσωπικό, triple. Πρόεδρε, συγγνώμη, με την 329 τι γίνεται, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θυμάτων. 29.01.01 29.01.01 ή 329 Θεωρήσουμε ότι καλύπτεται, λέει ο πρόεδρο. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Τρίπελ. Ξαναγυρίζω λοιπόν στο Insurance Against Sickness, ασφάλεια υγείας. Όλη η σελίδα αυτή καλύπτεται. Περνάμε στην επόμενη σελίδα. Καλύπτεται και αυτή εκτός της 4524 Ehrenhauser, αλλά είναι η ίδια πλειοψηφία εδώ. Περνάμε στην επόμενη σελίδα. 200 του αγγλικου 4552 ίδια πλειοψηφία. Και ερχόμαστε στο 20 λατινικό. Τι είναι, XX, χ είναι αυτό ή 20 λατινικό. Τι είναι. Πάση περιπτώσει, μετά είναι το 010101. Λίγο ο James Bond θυμίζει αυτό. Δαπάνε για το προσωπικό σε ενεργή δράση στα θεσμικά όργανα. Γιατί υπάρχει προσωπικό με ενεργή δράση, απασχόληση στα όργανα. Λοιπόν, μου λένε εδώ ότι 31-32 καλύπτεται. Αντίθετα, πρόταση της εισηγήτριας χωριστή ψηφοφορία από το 536 εισηγήτρια. Δεν το θέλω εγώ αυτό, δεν το ζήτησα εγώ αυτό. Μια πολιτική ομάδα το ζήτησε. Γιατί στην τροπολογία αρχικά ήταν της του ΕΛΚ τροπολογία, υπάρχουν πέντε όροι για διαφορετικά αποθέματα η τροπολογία τα παίρνει όλα μαζί με. Εγώ είμαι υπέρ όλων, αλλά το αίτημα είναι να ψηφίσουμε τους όρους τους πέντε αυτούς χωριστά έναν έναν. Όλα αυτά είναι στο 536. Πρέπει να πάρουμε το κείμενο της τροπολογίας. που έχει πέντε παραγράφους και ψηφίζουμε χωριστά τις παραγράφους. Αυτό ζήτησε μία ομάδα, η πράσινη. Έτοιμοι. Καταλάβατε. Πρώτη παράγραφος. Υπέρ. Κατά. Τι να κάνουμε, θα ψηφίσουμε. Ηλεκτρονικά. Ψηφίσουμε. Ο συντονιστής του ΕΛΚ τηλεφωνάει για να πάρει οδηγίες. Τι θα, τι θα πει, πώς ψηφίσεις το ΕΛΚ. Εγώ ψήφισα λάθος γιατί η Ίγκη ήρθε κακός. Πέρας. 22 υπέρ, 21, 18 κατά, εγκρίθηκε η πρώτη παράγραφος. Παράγραφος 2. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγώ δεν ψηφίζω. Ψηφίστε παρακαλώ. Στοπ. 21 5 18 κατά ίδια πλειοψηφία. Τρίτη παράγραφος. Υπέρ με τα χέρια. Με τα χέρια τώρα. Υπέρ. Κατά. Α, είναι σαφές. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικά. Άλλαξε η πλειοψηφία εδώ. Σε αυτή την παράγραφο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. επιταχύνεται η διαδικασία. Γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά εν πάση Πέρασε. 19 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται και η τρίτη. Τέταρτη παράγραφος. Ψηφίζουμε. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρας. 19 υπέρ 21 κατά. Απορρίπτεται η τέταρτη. Πέμπτη παράγραφος. Η κυρία Γένσεν. Πού, πού είμαστε, πού είμαστε, γιατί, γιατί έχω μπερδευτεί. Είμαστε στην τελευταία παράγραφο των σχολείων της 536. Οι τρεις πρώτες παράγραφοι εγκρίθηκαν, η τέταρτη απερίφθη, ψηφίζουμε την πέμπτη και τελευταία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. 19 πέρα 21 κατά. Απορρίπτονται και αυτοί. Στα σχόλια λοιπόν εγκρίνονται τρεις πρώτες παράγραφοι, οι άλλες δύο απορρίπτονται. Και εδώ ένα επιφανές πρώην μέλος και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου ήρθε όχι για να ψηφίσει, δυστυχώς, αλλά για να δείξει το ενδιαφέρον που απορρίπτει στις εργασίες της Επιτροπής μας. Να θεωρήσουμε οι 555 καλύπτεται. Δυστυχώς όχι. Και εδώ έχουμε πολλές ε, τροπολογίες. Όχι, όχι, μία. Μία. Για να μπει στο αποθεματικό. Η συγγήτρια υπέρ. Ηλεκτρονικά. 555. Η συγγήτρια υπέρ. Ψηφίζουμε. Πέρασε. 22 υπέρ, 18 κατά. Η υπόλοιπη σελίδα καλύπτεται. Διακόσα είναι το αγγλικό κειμένο. Καλύπτεται. 202. Πάμε στην 537, οι άλλες καλύπτονται και εδώ είναι για αποθεματικό, η λογική θα έλεγε ότι 537 θα πρέπει να έχει την ίδια μοίρα που έχουν και οι προηγούμενες. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξετε γνώμη. 537. Επειδή σε μια σελίδα μου φαίνεται. Όχι. Ναι, ναι, βιάστηκα, βιάστηκα λέει πρόεδρος. Έχουμε τροπολογία 5.36, αλλά σε διαφορετική γραμμή. Και 5.55 εδώ είναι όμως άλλη γραμμή, remuneration allowances, δηλαδή μισθοί και επιδόματα. Εγώ υποθέτω ότι καλύπτεται από την, από την ψήφο που κάναμε. Όχι, όχι, για μα πει η συγγετρία. Γυρίζουμε στο χ, χ, 01, 01, 01, 01, φορές 01, 536, 555, τι λέει η συγγετρία. Το τελευταίο 01 κάνει τη διαφορά. Γιατί αυτό που ψηφίσαμε πριν ήταν η επικεφαλίδα, ο τίτλος Τώρα μπαίνουμε σε υπότιτλους. Και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε τα νούμερα. Φαίνεται επανάληψη, αλλά δεν είναι. Γιατί 010101 για την 536 πρέπει να ψηφίσουμε ένα ποσό θα πρέπει να κάνω προφορική τροπολογία. Γιατί κάναμε χωριστή ψηφοφορία. Τρία στο παθηματικό εγκρίθηκαν και δύο απορρίφθηκαν. Πέντε εκατομμύρια απορρίφθηκαν. Πρέπει να τα βγάλουμε από το 12,5. Οπότε θα είναι 7,5 εκατομμύρια στο παθηματικό για την 536 και είμαι υπέρ του ποσού. Μία ψήφος δηλαδή εδώ. Μία ψηφοφορία. Η 536. Αλλά στο αποθυματικό όχι 12,5 εκατομμύρια αλλά 7,5 εκατομμύρια. ηλεκτρονικά Πέρας. Με 22-16 εγκρίνεται. 5 5-55 εισηγήτρια. Την ψηφίζουμε εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι υπέρ, τα χέρια. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρασε εγκρίνεται με 22-16. Κατ' επέκταση η υπόλοιπη σελίδα, σελίδα καλύπτεται. Γυρίζουμε σελίδα 01-02. Πάμε στην 537. Αποθεματικό. πληροφόρηση κλπ. Εδώ έχουμε σχόλια. Και στο κάτω μέρος της σελίδας, στη 01 02 01 στην 537 δηλαδή, έχουμε τα νούμερα. Ψηφίσουμε τις δύο ταυτόχρονα. Ωραία, ψηφίσουμε αυτές τις δύο τροπολογίες, 537 και τις δύο μαζί ηλεκτρονικά. Εισηγήτρια υπέρ. Πέρας. Απορρίπτεται με 19-20. Εισηγήτρια. Όχι, έχει 20, 20-20, πάλι απορρίπτεται. Υπάρχει και άλλη λύση. Να ψηφίσω εγώ στη θέση σας. Αν μου δώσετε εντολή, με την εντολή που θα δίνετε εσείς, αν θέλετε. Περνάμε στην επόμενη σελίδα. External Staff Working with Institution. Γυρίζω σελίδα. Contract staff. Καλύπτεται. National Civil Servants Temporary. Καλύπτεται. External staff. Το 3032 καλύπτεται. Η 520 όμως το ίδιο πρόβλημα. Δύο τροπολογίες 520. Η μία για τα σχόλια, η άλλη το νούμερο. Η συγγήτρια υπέρ. Ψηφίζουμε. ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται με 19-20. Ή 520. 31, 32 και 33 καλύπτονται. 259 ψηφίζεται. Η Η για την απελευθέρωση του αποθυματικού. Η συγκίτρια υπέρ. Υπέρ. Γκέραν φέρμα. Γιατί ποσό ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 259. Το νούμερο είναι 4 εκατομμύρια στο αποθεματικό. Και ψηφίζουμε και τα σχόλια, τους όρους κάτω του οποίους θα απελευθερωθεί το αποθεματικό. Δεν ψηφίζουμε νούμερα.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 Δεν ξέρω σε σχέση με τι άλλε ομάδε, αλλά είναι μια πολιτικά σημαντική τροπολογία για τον, την συναλλαγή, φόρο επί των συναλλαγών. Δεν λέει τίποτα άλλο σε σχέση με προσυπόμνηση, αλλά προετοιμάζει τη συζήτηση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα του φόρου ή τελου επί των συναλλαγών. Τώρα σε σχέση με τη συζήτηση υπό την Βελγική Προεδρία και για την λέσχη των 20 θα ήταν πολιτικά σημαντικό να τεθεί στο τραπέζι αυτό και γι' αυτό θέλουμε να υπάρξει αυτό. Δεν είναι κανένα πρόβλημα να το ψηφίσουμε τώρα. Αν θέλετε όμως ως τελικό στοιχείο που θα συμπεριληφθεί να ψηφιστεί πάλι συμφωνούμε. Η πρότασή μου είναι μάλλον να το, κρατήσουμε ε, για την τελική ε, διαπραγμάτευση γιατί αυτό που μας σήμισε ο Γκέραν Φέρν είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κρίμα τώρα να γίνει μια συζήτηση επί της ουσίας του σημείου αυτό. Προτείνω λοιπόν να μην το ψηφίσουμε αλλά θα το υποβάλουμε προς ψηφοφορία όταν θα υπάρξει γενική συμφωνία. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ψηφιστεί τώρα. Ο κύριος Σαλβαντόρ. Το ΕΛΚ έχει θέση για αυτή την τροπολογία και τώρα όπως και στην τελική συζήτηση θέλουμε να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία για αυτό το σημείο. Αλλά δεν έχουμε κάποια προτίμηση για τώρα ή στερότερα. Αλλά θα πρέπει να ψηφιστεί ξεχωριστά οπωσδήποτε. Donc je vais Οπότε θα χρησιμοποιήσω την εξουσία μου σαν Προέδρου και θα αρνηθώ να υποβάλω προς ψήφιση αυτή την τροπολογία. Κάποια στιγμή θα υποβληθεί. Πιστεύω όμως ότι εφόσον εδώ βρισκόμαστε σε μία πρόταση η οποία έχει μεγάλη πολιτική ε, σημασία που θέτει και νομικά και πολιτικά προβλήματα και πρέπει να εξεταστεί στα πλαίσια της διαπραγματεύσεως του πακέτου που θα προβληθεί στην ε, Ολομέλη μετά από τις συζητήσεις με το Συμβούλιο Υπουργών πιστεύω ότι θα επιφυλαχθούμε. Άρα τώρα δεν θα την ψηφίσουμε. Τελειώσαμε λοιπόν με την κατηγορία 5. του τμήματος 3 βέβαια της, της Επιτροπής. Και πάλι όμως βγάζουμε ένα αναστεναγμό ανακούφισης και θέλουμε ε, να δώσουμε τα πρώτα συγχαρητήρια στον εισηγητή, να ευχαριστήσουμε τα μέλη και για να μην χάνουμε το ρυθμό μας εξετάζουμε τις ε, γραμμές των άλλων θεσμικών οργάνων. Εάν λοιπόν η συγγήτρια των άλλων θεσμικών οργάνων, η κυρία Helga Τρίπελ, είναι έτοιμη. Λοιπόν, στο αγγλικό κείμενο και πάλι οι ίδιες τροπολογίες είναι και είμαστε στη σελίδα 210 στο αγγλικό κείμενο. Ο, η γενική επικεφαλίδα είναι Parliament Κοινοβούλιο και ξεκινάμε με τη γραμμή 1004 τακτικά έξοδα ταξιδίου. Θα ξαναβρεθούμε λοιπόν πάλι στις τροπολογίες του κυρίου Έρενχάουζερ να μειωθεί αυτή τη φορά κατά 15% το σύνολο των γραμμών Οπότε λέω να κάνουμε ό,τι κάναμε για την Γαλλία 5 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχήν να ψηφίσουμε ε, επί της αρχής αυτή την τροπολογία και να θεωρήσουμε ότι θα ισχύσει η ίδια πλειοψηφία για την ίδια κατηγορία τροπολογιών. Διότι μπορεί ο κύριος Αρενχάουζερ να έχει κάνει και διαφορετικές τροπολογίες, οπότε θα τις εξετάσουμε κατά περίπτωση. Λοιπόν, η 46 4619 τροπολογία του κυρίου Έρενχάουζερ υποβάλλεται προς ψήφιση ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η, ε, η τροπολογία 2002 της κυρίας Τρίπελ, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, ομόφωνα και ε, χαιρετίζω, συγχαίρω την εισηγήτρια. Η 41-28 ίδια πλειοψηφία, 41-11 ε, του κυρίου Χάρτογκ. Ε, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ο κύριος Χάρτονγκ λοιπόν έχει επίσης πολλές τροπολογίες που αναφέρονται σε μία διαγραφή των γραμμών οπότε και εκεί θα θεωρήσουμε ότι ισχύει η ίδια πλειοψηφία αν δεν έχει ταντήρηση. Αυτό ισχύει για το 41-12 το 41-12 του 1090-1091 ε, στο, στην επόμενη σελίδα έχουμε την ε, τροπολογία 20.009 της κυρίας Τρύπελ. ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές κανείς δεν είναι κατά άρα υιοθετείται η τροπολογία 20.01 της κυρίας Τρούπελ. ποιος είναι υπέρ 2001 της κυρίας τρύπελ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ο διά, διάφοροι συνάδελφοι από το Λουξεμβούργο θα χαρούν. Τώρα περνάμε στο κεφάλαιο 12.00. Ε, η τροπολογία 20.09 της κυρίας τρύπελ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 20.01 της κυρία Τρίπελ υπέρ ο εισηγητής είναι κατά ποιος είναι κατά Πολλοί. ποιοι απέχουν απορρίπτεται ομόφωνα τροπολογία 2010 η εισηγήτρια είναι κατά ποιος είναι υπέρ κατά αποχές επίσης απολύπτεται. Υπάρχει μια συμβιβαστική τροπολογία, λέει η κυρία Τρίπερ, και το 4208 για την 4208. Όχι, όχι. Υπάρχει... Ε, υπάρχει σε ένα άλλο έγγραφο η συμβιβαστική τροπολογία 42052. είναι το έγγραφο που ξεκινά με τροπολογία 2051. Όντως, έχουμε ε, χωριστά τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Οπότε, Εδώ υπάρχουν 7 τροπολογίες, 20, 51, 20, 52, 20, 54, 55 και 56 και 22, 51. Όλες βρίσκονται σε αυτό το τεύχος. Η κυρία Τρίπελ έχει τα ίδια έγγραφα. είναι πιο εύκολο ίσως να ψηφίσουμε πρώτα τις συμβιβαστικές τροπολογίες και μετά τις υπόλοιπες. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε όλες μαζί τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Μάλιστα. James. Θα ήταν χρήσιμο να τις παίρναμε μία προς μία τις τροπολογίες. Ιδιαίτερα στην 255 έχουμε όλα τα χρήματα ως κονδύλιο για τον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ήταν μια συνεδρίαση που έγινε σήμερα. Νομίζω θα πρέπει να έχουμε κάποιες αποσαφηνήσεις για το τι σημαίνει αυτό προτού προχωρήσουμε και εγκρίνουμε κονδύλιο τέτοια μορφή. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε χωριστά το 20-55 ε, ε, και οι άλλες όλες μαζί. Λοιπόν, ψηφίζουμε καταρχήν το 20-055. Ε, Ποιος είναι υπέρ. Ο εισηγητής είναι υπέρ και το ΕΛΚ είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Ε, αποχές. Υιοθετείτε όλες οι άλλες μαζί. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Όλες λοιπόν αυτές οι συμβασικές τροπολογίες θα μας ε, διευκολύνουν πολύ τη ζωή και επανερχόμαστε τώρα στο τεύχος με τις τροπολογίες το 4208 και το 605 καταπίπτουν γιατί είναι καλυμμένα η τροπολογία χάρτων 41-13 είναι η ίδια πλειοψηφία όπως και προηγουμένως. Το 2012 καλύπτεται. Πρέπει να το ψηφίσουμε. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το 42-09 καλύπτεται, το 4114 επίσης, το 566 επίσης, το 4115 και 35 είναι οι τροπολογίες χάρτων τις οποίες έχουμε ουσιαστικά καλύψει. Το 4318 καλύπτεται, όχι, είναι ζητά να το ψηφίσουμε. Συμφωνώ αν αλλάξουμε τα σχόλια και διαγράψουμε έτσι ώστε να μπορέσει να διαγράψουμε θεσμοί, θεσμικά όργανα σε σχέση με γλωσσικά μαθήματα ώστε τα, οι παρατηρήσεις ε, κατά τη διάρκεια δηλαδή των ε, ορών εργασίας να διαγραφούν. Sur Ίγκη ζητά να ψηφίσουμε τη, τα σχόλια. Τι, τι πιστεύει η συγκίτρια, είναι υπέρ? Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά σχετικά με αυτή την τροπολογία. Πρέπει να ξεκινήσουμε την, ε, ε, την ε, ψηφοφορία. Από πλευράς ΕΛΚ μπορούν να ψηφίσουν όλοι. Λίγη ψηφοφορία. 20 υπέρ 18 κατά, άρα εγκρίνεται η τροπολογία. Τώρα social welfare 608. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος σου είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Ε, μία μικρή πλειοψηφία υπέρ το 2003 για την κινητικότητα. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 41.16 και 41 και 40 είναι του κυρίου Χάρτονγκ, η ίδια πλειοψηφία δηλαδή. Το 20.08 είναι της εισηγήτριας η οποία αντιτίθεται καλύπτεται από τη συμβιβαστική. Μου λέγουν όχι. Είναι το contingency reserve και μου λέγουν ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Προτείνουμε να αφήσουμε το ίδιο ποσό όπως στις εκτιμήσεις. Εννοείται για το 2008. Ε, ναι και στις ε, ε, δύο τροπολογίες να κρατήσουμε τους αριθμούς των ε, ε, υπολογισμών, των υποθέσεων. 20.08 λοιπόν, κανείς δεν είναι υπέρ, όλοι είναι κατά. Ποιος είναι αποχή, κανείς. Απορρίπτεται. Το 563. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Επίσης απορρίπτεται. Enlargement Reserve. 20-12 τροπολογία της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46-29 Ερενχάουζερ είναι από αυτά που είπαμε η ίδια, η ίδια πλειοψηφία και τώρα είμαστε στο 2013 του εισηγητή Other Specific Property Management Arrangement ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το 564 της ομάδος ΕΛΚ. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το 2026 κεφάλαιο. Η συγγήτρια προτείνει καταρχήν να ψηφίσουμε την τροπολογία 568. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα οι άλλες καταπίπτουν. Δηλαδή οι 20.09 46-44 απορρίπτονται. Το, η 607 των πρασίνων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την 607 πάλι των πρασίνων. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έπιπλα 20.04 η είναι κατά ποιος είναι υπέρ κατά αποχές μόνο οι σοσιαλιστές στηρίζουν στην ίδια γραμμή Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αποσύρουμε την 570. Άρα δεν έχουμε τροπολογία σχετικά με ε, το, τα έπιπλα. 571. Τεχνικός εξοπλισμός. Το ΕΛΚ επιμένει στην τροπολογία της. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, οχήματα. Έχουμε μία τροπολογία 431 εισηγήτρια είναι κατά ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για τις τηλεπικοινωνίες η μία ομάδα έχει μία τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται όσον αφορά τις μετακομίσεις 20.05 ε, της ηγήτριας ποιος είναι υπέρ κατά αποχές άρα τα removals οι μετακομίσεις ε, εγκρίνονται δεν ξέρω αν θα μετακομίζουμε για να πάμε στο Στρασβούργο ή στις Βρυξέλλες τώρα ε, η 4637 του κυρίου Έρεν Χάουζερ είναι συνήθις άρα απορρίπτεται το 489 των ε, συντηρητικών ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4634 είναι μία η κυρία Γένσεν σχετικά με την διασκέδαση Φυσικά εδώ θα θέλαμε ο κύριος Μπούσεκ να μας έδινε ακόμα και σαμπάνια και στρίδια όλα αυτά θετικά θα θέλαμε υπεψηφιστή λοιπόν και υποστηρίζουμε αυτήν την τροπολογία. Ευχαριστώ. Είναι απόλυτα νόμιμο οι φιλελεύθεροι συμφωνούν με το 46-34 δηλαδή να μειωθούν τα θεάματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή έχουμε αρκετό θέαμα στην Επιτροπή Προπολογισμού δεν χρειαζόμαστε άλλο η 490 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές οι σοσιαλιστές θαραλέα απέχουν ή τουλάχιστον μία, ένα μέρος της ομάδας σοσιαλιστών διότι η Γιούτα Χάου δεν συμφωνεί. Περνάμε τώρα στην ε, Συν 490. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Η ίδια, για τους ίδιους λόγους. Τώρα στη γραμμή 3048, 2014 της ΕΛΓΑ. Μόνο σχόλια. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές το 2014 υιοθετείται. Μετά η γραμμή 3041 Expenditure on Travel Agency Services η 2006 της έργα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 19 λοιπόν υπερψηφίζεται Υπάρχει μη, ένα συμβιβασμός για τη γραμμή 320 για την τροπολογία 565. Μου λέγουν ότι υπάρχουν ε, παρατηρήσεις για το 606. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Έχουμε ψηφίσει το House of European History γιατί ο James ζήτησε χωριστή ψηφοφορία. Την 485 πρέπει να ψηφίσουμε τις παρατηρήσεις μόνο, τα σχόλια μόνο. Pardon, James. Ε, this is, uh... Αυτή είναι μια τροπολογία που συνδέεται σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο είχαμε ψηφίσει όσον αφορά το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε σχέση με το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια συνεισφορά σε σχέση με αυτό το πιλωτικό σχέδιο. Δεν είναι μια γραμμή που έχει χρησιμοποιείται και θα ήθελα να ζητήσω να υποστηρίξω. Euh, James parle du 485. D'accord. OK. Très bien. Donc, les deux premiers amendements. Là, για το 385. Λοιπόν, τώρα θέτουμε προ ψηφοφορία το 485 που εξήγησε ο Τζέιμ. Ο εισηγητή είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχέ. Δυστυχώ, απορρίπτεται. Περνάμε στο 32-42. Η 20-15 της Έργα Τρούπερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 486 ε, πρέπει να ψηφιστεί. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στο κέντρο ε, επισκεπτών. Τρεις τροπολογίες. 20.07 σχετικά με τον αριθμό της Έλγα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται. Το 2016. Σχόλια. Μόνο τα σχόλια. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 41-20 είναι η συνήθις τροπολογία του κυρίου Χάρτονγκ η οποία απορρίπτεται. Το επόμενο, 2017, μόνο το σχόλιο της Έλγα Τρύπερ. ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, ομόφωνα. Περνάμε εις ε, την ε, κοινοβουλευτική τηλεόραση, Web TV, το 4121 και το 4643 Νομίζω ότι όλη η γραμμή καλύπτεται από τη συμβιβαστική λύση. Ο κύριος Χάρτονγκ θέλει κάτι να μας πει. Θα ήθελα να ψηφίσουμε αυτήν την 4-1-2-1 αν γίνεται. Να την ψηφίσουμε. Uh, Ευχαρίστω, αλλά μου λέγουν ότι ε, ο συμβιβασμός ε, καλύπτει το, την τροπολογία αυτή. Αλλά αν θέλετε να ψηφιστεί, τι να κάνουμε. Λοιπόν, 41-21, ποιος είναι υπέρ. Ε, υποθέτω ότι ο κύριος Σαρτόγκ είναι υπέρ της τροπολογίας του. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απερίφθη λοιπόν η τροπολογία και είχε υπερκαλυφθεί ήδη και οι υπόλοιπε στην ίδια γραμμή είναι υπερκαλυμμένες. Ο κύριος Φερνάντσο έχει μία παρατήρηση για το 659 να το αποσύρουμε. Το 487 όμως διατηρείται, οπότε ψηφίζουμε, ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ της 487. Ε, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 4350. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. όχι μόνο όμως βλέπω περίεργους ε, συμμαχίες. Οπότε ηλεκτρονική ψηφοφορία ξεκινά. Για το 4350 ε, θα, θα ψηφίσω γιατί δεν έχουμε αρκετούς ΕΛΚ. Θα προσθέσουμε και την συντονία που είναι αντίθετη. 31 κατά και 7 υπέρ. Είχα δει πάνω από 7 που είχα σηκώσει το χέρι προηγουμένως. Α σημειώνουμε όμως ότι η 4350 κατεψηφίσει. Η ε, 2018 της ΕΛΓΑ, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά έχουμε τις δύο του κυρίου Χάρτον Χέρενχάουζεν που έχουν την ε, ίδια αντίθετη ε, πλειοψηφία και ε, περνάμε εις το Parliamentary Assistance 2011 του εισηγητή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 46 17 είναι διαφορετική από τις συνηθισμένες. Μάλλον είναι ταυτόσιμη, συγχωρείτε. Όχι, δεν είναι ταυτόσιμη. Πρέπει λοιπόν να ψηφιστεί η 46-17 του κυρίου Ερενχάουζερ. Ποιος είναι υπέρ, ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι κατά, αποχές, απορρίπτεται η 499 των ε, συντηρητικών. Ο εισηγητής είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. Αποχές απορρίπτεται. Η 653 των ε, φιλελευθέρων και δημοκρατών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Και οι δύο μεγάλες ομάδες. Άρα έχασε και η επόμενη καλύπτεται και όλες αυτές απορρίπτονται. Πηγαίνουμε τώρα στο ε, δικαστήριο. Με συγχωρείτε, λέει. Ναι, ναι, ναι, είχα αφαιρέσει το Συμβούλιο, αλλά το Συμβούλιο χρειάζεται χρήματα sur Κάμε το Συμβούλιο, μπορούμε να τα ψηφίσουμε όλα μαζί εφόσον είναι ο ίδιος συντάκτης και το ίδιο πνεύμα. Ποιος είναι υπέρ του, ε, της τροπολογίας Χάουζερ για το Συμβούλιο. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται όλες. <coughs> Πάει το Συμβούλιο. Περνάμε στο δικαστήριο. 22.00. Καλύπτεται. 42.03 καλύπτεται. 42.00 καλύπτεται. Ε, συγγνώμη, 22.00 καλύπτεται. 42.03 καλύπτεται. 22.00 temporary allowances καλύπτεται. 42.03 πλειοψηφία κατά. Συντάξεις 22.00. 42.03 επίσης πλειοψηφία κατά. Αποστολές 42.03 πλειοψηφία κατά. 45.19 πλειοψηφία κατά. Training 42.03 πλειοψηφία κατά. Provisional Appropriation 42.00 καλύπτεται 42.03 πλειοψηφία κατά officials and temporary staff. 22.07 θα την ψηφίσουμε. Η άλλη είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Τρει, τέσσερι αποχε Εγκρίνεται. 120. Μισθή και άλλα δικαιώματα. Καλύπτεται. Συμβαστική 2251 το κάλυψε, το κάλυψε. Την 2201. Πρέπει να ψηφίσουμε την 2206. Είναι θέσεις για την Κροατία στο αποθεματικό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Γυρίζω σελίδα 12.00 αμοιβέ και επιδόματα 22.00 καλύπτεται 22.01 και αυτή ψηφίζουμε την 22.06 Κροατία αν είχαμε μια τροπολογία να καλύπτει όλα τα της Κροατίας δεν έχουμε από ξαναδώ τη λέξη Κροατία θα θεωρήσω την ίδια πλειοψηφία. Εξώ να βγει Σλοβαίνο και πει ότι εγώ δεν συμφωνώ. 22-06 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 42-03 καταπίπτει. 142 καλύπτεται. Υπερορίας πληρωνόμενες. Οι συνεργάτε τη Επιτροπή μα πολλέ φορέ κάνουν υπερορίε. 22.00 καλύπτεται. 42.03 πλειοψηφία κατά. 12.04 τα δικαιώματα με την είσοδο στην υπηρεσία και αποχώρηση από την υπηρεσία. 22.00 καλύπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε την 22.02. Εισηγήτρια. Υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 42.03 πλειοψηφία κατά, 143 καλύπτεται. 12.20 42.03 σαρανταδύμιδεν Άρτογκ, πλειοψηφία κατά, 129, προσωρινές πιστώσεις, 22.00 καλύπτεται, 22.03, συμβαστική για 29 νέες θέσεις. Ψηφίζουμε. Εισηγήτρια υπέρ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Οι άλλες δύο καταβίπτουν. υπό προσωπικό 22.00 καλύπτεται. 42.03 πλειοψηφία κατά. Το ίδιο εκεί 4203 από κάτω. Το ίδιο και για την γραμμή 1405 και για την 1406. Γύρισε σελίδα. 149. Provisional Appropriation. 22.00. Καλύπτεται. 4203 επίσης. Το ίδιο 1610, 1612, 162 αποστολές. 1630 κοινωνικά επιδόματα. 1632, 1650, 1654, 200. Η τροπολογία 2204 τρίπελ. Ψηφίζουμε την 22.04 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η άλλη είναι ταυτόσιμη. 21.02. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η άλλη είναι ταυτόσιμη. Για το ελεγκτικό συνέδριο όλα καλύπτονται. Αποστολές επίσης όλα τα από κάτω τροπολογή Ερενχάουζερ η πλειοψηφία κατά το ελεκτικό συνέδριο θα έχει πολλά λεφτά, θα πρέπει να είναι ευχαριστημένο. Η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή 814, 804 συγγνώμη των Σοσιαλιστών Αποσύρθηκε, μάλιστα. 804 αποσύρθηκε. 1004 επιδόματα οδηπορικά και ταξιδίου κλπ. Οι 2400 της Έλγκας ψηφίζεται υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Οι άλλες δύο καταπίπτων. 1008 και εδώ είναι οδηπορικά κοινωνικο-οικονομική. Οι σοσιαλιστές αποσύρουν την τροπολογία. Και το ίδιο και η 105 αποσύρθηκε. Κατά τους σοσιαλιστές δεν χρειάζεται ούτε οδηπορικά, ούτε άλλο τέτοιο είδους επιδόματα, ούτε κατάσταση, ούτε εκπαίδευση, Το γλώσσες η Οικονομική και η Οικονομική Επιτροπή. Μας απλοποιείται την κατάσταση. Ε, μόνιμη και προσωρινή η Τροπολογία 2401 της ΕΛΓΑ. Ψηφίζουμε. 2401. Κατά. Ευχαριστώ. Εγκρίθηκε. 2403. Θέση που σχέση με τη Λισαβόνα. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 1200 αμοιβές μισθή. 2.402 ψηφίζουμε. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 24.03 Λισαβόνα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε με την ίδια πλειοψηφία. 2.404 καλύπτεται. 42.04 Χάρτον το ίδιο. 785 καλύπτεται. 807 επίσης. 2403. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129. 2402. Έλεγα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2403 έλγα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Υπό προσωπικό 2405 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42.04 απορρίπτεται 24.05 της Χέλγα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περαιτέρω τις σοσιαλιστές αποσύρουν την 8.14 δεπάνες αποστολών σοσιαλιστές την αποσύρουν 2001 Χάρτον Ξέρουμε το αποτέλεσμα. 2007 ψηφίζουμε. Υπέρ, τροπολογία τρίπελ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24.07 της Χέλγα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 2.100. 24.06 της Χέλγα για τις 11 ε, νέες θέσεις υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 2408 της Χέλγκα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 808 δεν είχαν καν το χρόνο την αποσύρουν στους ελληνιστές, και είχε εξαφανιστεί. Τηλεπικοινωνίες 2408 Χέλγα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 816 αποσύρεται 809 καλύπτεται περνάμε στο επίπλωση 2410 εδώ είναι οι καρέκλες που θα καθίσουν οι 11 νέοι υπάλληλοι υπέρ κατά αποχές. Η κυρία Άντρας δεν θέλει τα νέα μέλη να κάθονται, να μην έχουν καρέκλες. Κάνει γυμναστική. Εγκρίθηκε η τροπολογία. 813 καταπίπτει, 214. Η 2408. έργα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 805 αποσύρεται ή 8 ή εκεί 815, 2548 τροπολογία χάτων την ξέρουμε, 810 σοσιαλιστές αποσύρεται, όχι όχι, α, 810 ψηφίζουμε, η συγκίτρια είναι υπέρ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 802 επικοινωνία. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Είναι κατά, κατά. Όχι, έχει λάθος. Αποσύρθηκε αυτή η 802. Επιτροπή Περιφερειών Τροπολογία Τρίπελ για τις συνεδριάσεις του Προεδρείου για τις Ολομέλειας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η επόμενη καλύπτεται. 12. 25.04. Της Χέλγα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25.00 παρατηρήσεις της Χέλγα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μισθή. 25.03 της Χέλγα και εδώ σχέση με τη Λισαβόνα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Χίλια διακόσα μισθή και επιδόματα 25.01 καλύπτεται. 25.03 ψηφίζουμε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 25.04 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 41.97 Χάρτον, ξέρουμε το αποτέλεσμα. 736 αποσύρεται. Καλύπτεται. 737 καλύπτεται. 783 επίσης. 1204. 2505. Της Για τις νέες θέσεις. Περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 818 καταπίπτει. 129, 2506, Χέλγα. 18 θέση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 καταπίπτει. Λοιπόν προσωπικό. Η πρώτη καλύπτεται, η μόνη που θα ψηφίσουμε είναι η δεύτερη, 2507 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι άλλες καλύπτονται. Δεκατέσσερα Θερμηνία. 25.08 της Χέλγκα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 740 καλύπτεται. 1404, 2509, Χέλγα. Εθνική Εμπειρογνώμη, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 741 κατά πίπτη. 1420-2510 της Χέλγα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 742 πίπτη. περιτερω Περιτέρω κατάρτιση. 25-11 χέλγα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 742 καταπιπτει πίπτη. 41-99 χάρτον γνωστή. Απορρίπτεται δηλαδή. 21-02, 25-12, χέλγα. Ε, ε, ηλεκτρονικό για υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε 25, 12, κατεπίπτει 744, έπιπλα, 25, 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε 745, καταπίπτει, 25, 14, χέργα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 746, κατά καταπίπτει, παρατηρητές. 25-15. έλεγα Πάλι οι Κροάτες εδώ. Παρατηρητές τώρα. Και όπως με εδώ ψιθυρίζει ο γραμματέας πρέπει να μπουν στο αποθεματικό. Τη μέρα βέβαια που οι παρατηρητές θα έρθουν στο κοινοβούλιο έρεται η απαγόρευση του αποθεματικού. Υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίθηκε 2516 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 47 πίπτη καταπίπτει 2-600 τροπολογία Το έλεγε κοιμάται. Θα ψηφίσουμε ρήμην του. Κατά αποχές εγκρίθηκε 25-17-7-48 κατά πίπτη. Ο διαμεσολαβητής 26-01 Χέλγα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τα υπόλοιπα καλύπτονται 100 και 103 για το λαβητή. Οι 1200 επίσης 1400 επίσης Οι 231 έχουμε τροπολογία 5 Χάρτογκ να καταργηθούν τα κονδύλια αλλά ξέρουμε τι τύχη θα έχει αυτή η τροπολογία 1000 σοσιαλιστές την αποσύρουν. 110 πρέπει να ψηφίσουμε την 2701. Έλγα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1100. Η πρώτη τροπολογία καλύπτεται. 2701 για δύο θέσεις. Αυτό είναι το European Data Protection Supervisor. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι άλλες τρεις καλύπτονται. 2013. 4201 χάρτο. καταγύριζε σελίδα και τι βλέπω δεν έχω σελίδα. Όμως Υπάρχει ένα όμως. Υπάρχει ένα όμως έλεγα. Δεν τελειώσαμε. Θα τελειώσουμε με δύο ε, τροπολογίες που σας μοιράστηκαν σε δύο χωριστά φύλλα. που είναι για το τμήμα 10, ένα νέο τμήμα του προπολογισμού που δημιουργούμε, για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Έχουμε δύο τροπολογίες εδώ. Δεν μοιράστηκαν. Για να δούμε τις πήρατε ή όχι. Μοιράστηκαν στην αρχή, αλλά είχαμε τόσο πολλά χαρτιά που μάλλον ορισμένοι χάσαν τα χαρτιά τους. Ε, αντιπρόεδρε, μάλλον Δύο τροπολογίες σας έλεγα λοιπόν. Δεν ξέρω ποιος πρότεινε, η Έλγα, η Συντόνια, κάποιος να μας εξηγήσει με δύο λόγια τι λένε αυτές τις τροπολογίες και προτείνω να ψηφίσουμε ένα μπλοκ και τις δύο μαζί. Ποιος από τις δύο, ποιος, ποια θα μας φασίσετε. συνταγή. Προσπαθήσω να εξηγήσω. Αυτές οι δύο τροπολογίες που πήρατε συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Διπλωματική Υπηρεσία, Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Μία από αυτές είναι κοινή τροπολογία σε σχέση με το τμήμα 3 και το 10 που επεξηγείται επίσης και στον τίτλο και αυτή η τροπολογία ακολουθεί το αίτημα της ΑΦΕΤ Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και είναι μια τροπολογία στο 1901 0101 κονδύλιο για ανθρωπιστικές ε, δράσεις. Είναι μια γραμμή που συνδέεται με δαπάνες για τα στελέχη όσον αφορά την Γενική Διεύθυνση για την Εξωτερική Διπλωματική Δράση. Αυτή η τροπολογία είναι μια τροπολογία που δημιουργεί ένα αποθεματικό που συνδέεται στις δικές μας προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποβληθεί μια πρόταση για την μετάθεση στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Γενική Διεύθυνση, από τη Γενική Διεύθυνση ΡΕΛΕΞ για την εξωτερική υπηρεσία, την διπλωματική υπηρεσία για την δημιουργία μέτρων ειρήνευσης και αντιμετώπισης κρίσεων τι από πλευρά των συναδέφων τη ΑΦΕΤ αυτό αναφέρεται σε σχέση με δεσμεύσει που έγιναν από πλευρά τη ΥΠΑ τη εκπροσώπου Λέδη Άστον. 1.374.000 ευρώ είναι το κονδύλιο. Αυτό δεν προέρχεται από το πουθενά. Αυτό το κονδύλιο είναι μια κατεκτήμηση 70 στελεχών, 70 θέσεων κονδύλιο επίπεδο σε σχέση με την απασχόληση για ένα χρόνο αυτές οι, αυτές οι θέσεις. Συνιστώ να υπερψηφιστεί αυτή η τροπολογία που δίνει στο Κοινοβούλιο προφανώς να ξαναδεί την Λέδη Άστον και να το ξαναδεί το θέμα. Ευχαριστώ. Και το δεύτερο να εξηγήσω το δεύτερο. Euh, Έχω μία ερώτηση. Σε μια από τι τροπολογίες λέμε 18 νέε θέσει, στο όλοι 17 νέε θέσει. Λάφο. Προέβαινε, Λάθος είναι. Συντόνια. Πρόεδρε, εξήγησα τώρα μία από τις τροπολογίες. Υπάρχει και άλλη μία τροπολογία. Να συνεχίσω με την άλλη τροπολογία ή όχι. Η άλλη λοιπόν τροπολογία αφορά μόνο το τρίτο τμήμα, εξωτερική υπηρεσία, υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Ακολουθεί πάλι το αίτημα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Και η Χέργα Τρούπερ εγώ προτείνουμε να εγγραφεί στο αποθεματικό κονδύλιο που αφορά το υπαριθμόν 1, τον υπαριθμό 1 τροποποιητικό προϋπολογισμό και για το 2011 για τον προϋπολογισμό σε σχέση με την εξωτερική υπηρεσία και αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, διορθωτικό προϋπολογισμό 6, η κατεκτήμηση είναι 18,6 εκατομμύρια ευρώ και έχει ως εξής 5,3 εκατομμύρια στο γενικό επιτελείο και 13,3 εκατομμύρια σε σχέση με τις αντιπροσωπείες. Αυτή είναι η επεξήγηση. Η τροπολογία έχει ως εξής. Λέει, εγγράφει στο αποθεματικό 18,6 εκατομμύρια ευρώ από ένα συνολικό κονδύλιο για τους μισθούς συμπεριλαμβάνοντας και την διορθωτική επιστολή υπαριθμών 1 και τους όρους φυσικά οι όροι είναι ότι το αποθεματικό αυτό θα απελευθερωθεί μόλις η είπατη εκπρόσωπος η Λέδη Άστον ρητά και δεσμευθεί να διαβουλεύεται με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την στελέχωση των υπηρεσιών. Υπήρχαν κάποιες ανησυχίες που δημιουργήθηκαν στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τη στελέχωση της διπλωματικής υπηρεσίας. Σκέφτηκαν να εγγραφεί στο αποθεματικό για να υπάρξουν αποσαφηνίσεις από την κυρία Άστον. Συνιστώ να υπεψηφιστούν αυτά τα δύο. Ευχαριστώ. Merci. Alors, la Commission a demandé Ρωτήσω την Ίγκερ να μας πει και αυτή τη γνώμη της γιατί παρακολούθησε αυτές τις διαπραγματεύσεις για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και ψηφίσουμε την έκθεσή της στην αρχή για τον δημοσιονομικό κανονισμό και η Κομισιόν θα κάνει τη σχολιά της Πρόκειται για το μέσο σταθερότητας και για το θέμα αν το μέσο σταθερότητας που το Συμβούλιο το θεωρεί δικό του πεδίο ειδικά του χρήματα, αν αυτό θα είναι κοινοτικό όργανο ή αν θα δοθεί στα χέρια του Συμβουλίου. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση και χαίρομαι για το ότι οι αρμόδιοι για την εξωτερική πολιτική το έχουν αντιμετωπίσει με αυτό το θέμα. Το θέμα είναι εκείνοι που σχεδιάζουν, όχι προγραμματίζουν, σχεδιάζουν ένα μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσης δεν μπορεί να προγραμματίζεται, σχεδιάζεται. Θα παραμείνει υποκοινοτική επιρροή ή θα φύγει στα χέρια μιας μονάδας επί της οποίας εμείς δεν θα μπορούμε να έχουμε επιρροή μέσα στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής. Merci. Monsieur le directeur. Merci, Monsieur le Président. Uh, I, I just wanted to, to complete perhaps the, the, uh, the explanation on what it is about and the split of the uh, resources between what stays Η μονάδα αυτή τη στιγμή και τα άτομα που απασχολούνται ως επιτοπλίστων ασχολούνται με το να παρακολουθούν τα προγράμματα και τη συνέχεια δίνεται στα προγράμματα, την οικονομική συνέχεια που δίνεται, γιατί σας θυμίζω ότι την ευθύνη για την εφαρμογή του εργαλείου για την σταθερότητα της κοινή εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, την ευθύνη λέω, την έχει η Κομισιόν. Και γι' αυτό τα κονδύλια αυτά είναι στον προπολογισμό της Κομισιόν. Σας είπα, τα άτομα που ασχολούνται με αυτό ετοιμάζουν τις οικονομικές αποφάσεις που η Κομισιόν εγκρίνει και η Κομισιόν αναλαμβάνει την ευθύνη γι' αυτό. Η Κομισιόν δεν έχει βέβαια τα άτομα που θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τα προγράμματα αυτά. Αν, δεν τα εγκρίνεται θα είναι σαν να υπονομεύεται τη δυνατότητα δράσης της Κομισιόν για μια υγιή δημοσιονομική διαχείριση. Και σας θυμίζω επίσης την απόφαση του Συμβουλίου για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δίνει την ευθύνη στη νέα υπηρεσία για τα προγράμματα και για το εργαλείο σταθερότητας. Αυτά είναι εργαλεία γρήγορης δράσης σε περίπτωση κρίσης Οπότε πρέπει να εξασφαλιστεί μια ισορροπία ανάμεσα στον, στις απαιτήσει προγραμματισμού και στην πρακτική εφαρμογή μέσω των εργαλείων αυτών που επαναλαμβάνω είναι της ευθύνης της Κομισιόν. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά Σαφής. Ο κύριος Άλβαρο. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποσαφήνιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει πιο δύσκολη την απόφασή μου να ακολουθήσω ή όχι τη σύσταση τη εισηγήτρια, διότι κατανοώ τον λόγο πίσω από αυτό. Πρώτον, δεν είμαι μέλο τη επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είναι δύσκολο για μένα να γνωρίζω τι βρίσκεται πίσω από αυτό. Και για το δεύτερο το ίδιο, διότι αν διαβάσετε τους όρους απελευθέρωσης του αποθεματικού, μόλις η ύπατη εκπρόσωπος θα δεσμευτεί να διαβουλεύεται με το Κοινοβούλιο για τη στελέχωση της εξωτερικής υπηρεσίας ή θα έχουμε και δεν ξέρω πόσα και ποια στελέχη. Γενικά προτεραιότητες για στελέχη, κάνουμε λόγο για τις ε, ε, δυνατότητες που υπάρχουν τους καλύτερους ή για ίσονο σημασία θέσεις, θέσεις στελεχών. Δεν γνωρίζω για ποιο πράγμα γίνεται λόγος εδώ και αισθάνομαι ότι αυτό το πράγμα υπερβολικά βιαστικά ρυθμίζεται έτσι. Αν εσείς θεωρείτε ότι αυτό βαίνει καλό, σε έστω. Αλλά έχω κάποιες επιφυλάξεις. Το βρίσκω κάπως αξιοπερίεργο. Στο Ιούτα. Σύμφωνα με τις επεξηγήσεις, τις διευκρινήσεις που μας δόθηκαν και εγώ πιστεύω ότι εμείς δεν πρέπει να προδικάσουμε τίποτα και να μην βιαστούμε και στη δημοσιονομική μας διαδικασία εδώ. Πρέπει κάπως πιστεύω να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε περισσότερο τι πρέπει να γίνει σίγουρα κάποτε την εφαρμογή της διορθωτικής επιστολής πρέπει να την προωθήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει σε αυτή τη φάση να υποχωρήσουμε στα αιτήματα των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Μου φαίνεται κάτι υπερβολικά επικίνδυνο για αυτή τη στιγμή. Ας περιμένουμε, ας αναμείνουμε πρώτα, να μην χαλάσουμε, να μην κάνουμε καμιά ζημιά η Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων θα δημιουργηθεί οπωσδήποτε. Πώς όμως θα στελεχώνεται και από ποιο κονδύλιο θα τροφοδοτείτε, ίσως βιαζόμαστε υπερβολικά να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά τώρα. Οι διευκρινήσεις που μας δόθηκαν δεν σημαίνει να ε, αφήσουμε τα χέρια από αυτό. Ευχαριστώ. Ε, δεν ξέρω αν κάποιο άλλο είναι μέλο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εγώ είμαι μέλο. Σε αυτή τη φάση είναι σημαντικό, πιστεύω, να ακολουθήσουμε τα μέλη την, τη σύσταση των κοινοβουλευτικών επιτροπών σε σχέση με τις ε, δράσεις και να μην προσπαθούμε να μαντεύσουμε τι θέλει να κάνει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα για αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την υλοποίηση διαφορετικών αποφάσεων. Πρέπει να ακολουθήσουμε, θα έλεγα, τη σύσταση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σε αυτή τη φάση, στην πρώτη ανάγνωση. Και μετά μπορούμε να καταλήξουμε στη διαδικασία συμφιλίωση, συνδιαλλαγή. Α ακολουθήσουμε αυτή τη σύσταση Τη της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Και πρέπει να αποκαλούμε με συνέπεια το αξίωμα την ε, κυρία Άστον. Δηλαδή είπα το εκπρόσωπο ή αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Λέδη Άστον. Βαρώνη Άστον είναι το όνομά της. Αυτό θα ήταν ακριβέστερο. <laughs> Αντιλαμβανόμαστε αυτή την ε, προφορική τροπολογία. Η κυρία Νίνσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να βρίσκεται κανείς μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Η Χέλγα είχε δίκιο. Να περιμένουμε λίγο περισσότερο. Να δούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια από πού θα αντληθούν αυτά τα χρήματα, αυτό το κονδύλιο. Ίσως στις επόμενες εβδομάδες η κατάσταση θα είναι σαφέστερη. Φυσικά είναι και ένα θέμα χρόνου αυτό και δεν μπορούμε να περιμένουμε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως θα μπορούσα να συστήσω αύριο κατά τη διάρκεια συνάντησης των μελών της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων να γνωστοποιήσω τις επιφυλάξεις σας και να δούμε αν μπορούμε να συντονίσουμε μια κοινή θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και απευθύνουμε στους συντονιστές. Αντιλαμβάνουμε ότι διάφοροι ραμέλοι του ε, Προεδρείου έχουν θέσει τις αμφιβολίες τους και βεβαίως ε, ε, αναφερόμαστε στα μέλη μας, ε, τα εξαίρετα μέλη μας που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ιδίως τους Γερμανούς συναδέλφους, αλλά αυτή η διατύπωση είναι κάπως ομή. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσο δεν υπάρχουν ε, ε, περιορισμοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κρατήσουμε στο αποθεματικό τις πιστώσεις. Αυτό που προτείνω εγώ και εδώ επαφίεμαι στους συντονιστές είναι να μας δώσετε λίγο χρόνο. Δεν έχουμε υποχρέωση να το ψηφίσουμε αυτό απόψε. Έχουμε χρόνο μέχρι την Πέμπτη και για δύσκολες τροπολογίες που ε, θα περιληφθούν στην τελική πολιτική απόφαση απόφαση θα αποφασίσουμε 5 και 6 Οκτωβρίου. Είμαι λοιπόν της νόμης να μην τα ψηφίσουμε αμέσω, να τα συζητήσουμε όπως πρότεινε η Ναντέτζα με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, να δούμε τι γίνεται και αν διατηρήσουμε αυτές τις τροπολογίες να έχουμε κάποια διατύπωση η οποία να σέβεται περισσότερο τα άλλα θεσμικά όργανα και τους εκπροσώπους της. Συμφωνείτε να προχωρήσουμε έτσι. Το ΕΛΚ συμφωνεί με αυτή την άποψη. Ωραία. Οπότε δεν θα τα ψηφίσουμε και άρα αγαπητοί συνάδελφοι τελειώσαμε με τρία λεπτά, τρία λεπτά πριν τις 6.30. Ευχαριστώ τους δύο συγητές, όλα τα μέλη και σας δίνω ραντεβού αύριο σε 9 η ώρα το πρωί για να ξαναξεκινήσουμε αυτή την ε, αυτή τη συμφωνία και θα κρατήσω μόνο τους συντονιστές απλώς διακόπτεται η συνεδρίαση για λίγα λεπτά.